την καθυστέρηση των σημαντικών φορολογικών θεμάτων. Αυτό είναι το γενικό υπόβαθρο. Εκ μέρους του Sven Giegold παρουσιάζω την έκθεση για το πρόγραμμα Φισκάλης που προτίθεται να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να υπερβούν κάποιους φραγμούς προς όφελος των πολιτών τους. Το πρόγραμμα Φισκάλης είναι πολύ επιτυχημένο και δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που ξεκινούν από τη συνεργασία μεταξύ εθνικών φορολογικών αρχών. Από την θέσπιση του, το πρόγραμμα Φισκάλης διευκόλυνε και ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βοηθήσει τις εθνικές φορολογικές αρχές ε, να ε, ε, εκπληρώσουν το βασικό τους καθήκον της ίσφραξης φόρων. Η έκθεση έτυχε της ευρεία υποστήριξη πολλών πολιτικών ομάδων και χαίρομαι διότι η πλειοψηφία των βουλευτών αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας, αυξημένη συνεργασία στο φορολογικό τομέα και αύξηση του αντίστοιχου προπολογισμού. Μία τροπολογία μόνο έχει υποβληθεί για την αυριανή ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θέλουμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σα για την τροπολογία αυτή. Το μέσο των διασυνοριακών κοινών ελέγχων είναι το τελευταίο, ο τελευταίος φραγμός για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών διαφορετικών κρατών μελών. Η κοινή έλεγχη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις ε, του transfer pricing ε, και των επιθετικών φορολογικών σχεδιασμών. Σας παρακαλούμε λοιπόν να ψηφίσετε υπέρ της κοινή τροπολογίας σοσιαλιστών και πρασίνων ούτως ώστε η κοινή φορολογική έλεγχη να είναι επιλέξιμη βάσει του προγράμματος φυσκάλη. Αυτό θα επιτύχει δίκαιη φορολογία προς όφελος όλων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη Επιτροπής, το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Έτιγκερ. Äh, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ο συνάδελφος Μοσκοβισή βρίσκεται στην Αθήνα για συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση και τον εκπρόσωπο εγώ εδώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Σκοτ Κάτω ε, να μεταφέρει τους χαιρετισμούς μας στον συνάδελφο Σβέν Γκίγκολτ και να τον ευχαριστήσετε για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για το φάκελο αυτό. Όπως ε, και πριν, οι ε, εθνικές φορολογικές αρχές δεν έχουν επαρκή δυνατότητα για επαρκή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει και για τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Λόγω της έλλειψης συνεργασίας υπάρχει έλλειμμα στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη. Και θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις για την ψηφιοποίηση και τα νέα μοντέλα φορολογικής απάτης που μπορούν να σχεδιάζονται. Θέλουμε να απαλλάξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από περιτά φορολογικά βάρη. Αυτά τα περιτά φορολογικά βάρη επιβαρύνουν τις εθνικές φορολογικές αρχές. Οι εθνικές φορολογικές αρχές πρέπει να ασχοληθούν με το βασικό τους καθήκον, που είναι η ίσπραξη φόρων. Και αυτό θα είναι προς όφελος και των εθνικών και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα Φισκάλης αυτό το σκοπό έχει, να βοηθήσει τη συνεργασία των φορολογικών αρχών με μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την επιχειρησιακή συνεργασία των φορολογικών αρχών. Η συνεργασία θα συμπεριλαμβάνει και ε, πληροφοριακά συστήματα και ε, βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η σειρά μέτρων που προτείνονται θα βοηθήσουν την εσωτερική αγορά και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο πρόγραμμα Φισκάλης για τα έτη μετά το 2020 θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να επιτευχθεί φορολογική δικαιοσύνη. Ένα σημαντικός περαιτέρω στόχος ε, του προγράμματος φυσκάλης είναι το να διευκολύνει την εργασία των φορολογικών αρχών και να εξυγχρονίσει τη λειτουργία των ε, φορολογικών αρχών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το βάρος για τους φορολογουμένους. Έχει διάφορες συνιστώσεις το πρόγραμμα Φισκάλης. Βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών μέσω ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Δεύτερον, εισάγει καινοτομίε, για τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως τεχνολογία blockchain τρίτον βελτιώνει τον συντονισμό και με καινοτομίε πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών βελτιώνει τη συνεργασία των φορολογικών αρχών και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, καταρτίζοντας το προσωπικό και εκπαιδεύοντας ε, τους συνεργάτες. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να είναι σωστά ενημερωμένο το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Το πρόγραμμα Φισκάλης δεν είναι καινούριο. Το υφιστάμενο πρόγραμμα έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και στο παρελθόν. Υπάρχει προστιθέμενη αξία του προγράμματος για τις φορολογικές αρχές και χαίρει ιδιαίτερη εκτίμησης από τις φορολογικές αρχές. Οι κοινοί φορολογική έλεγχοι και οι κοινέ ομάδε εμπειρογνωμόνων χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Φισκάλη και για την επόμενη φορολογική περίοδο προβλέπονται 270 εκατομμύρια ευρώ. για τη βελτίωση της φορολογικής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι ένα εξυγχρονισμένο πρόγραμμα φυσκάλης θα είναι ε, υπέρ της φορολογικής συνεργασίας ε, και της βελτίωσης των φορολογικών υπηρεσιών. Και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έχει καταβληθεί σημαντική δουλειά για να προχωρήσει αυτό το θέμα και μέσω της δουλειάς του κυρίου Γκίγκολτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω επικοδομητικές συζητήσεις Και ε, να απαντήσω σε κάτι που ρωτήσατε στην αρχή, γιατί δεν βασιστήκαμε στο άρθρο 116 στην χθεσινή πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχει αρχή της πλειοψηφίας στα φορολογικά θέματα για να επιλέξουμε την ε, κατάλληλη οδό ε, για να περάσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Θα δώσει μικρότερο δικαίωμα εποπτείας στο Συμβούλιο ε, το άρθρο 116. Ο κύριος Μουσκοβισή, συναδελφός μου, τις επόμενες εβδομάδες θα έχει την ευκαιρία να το συζητήσει περισσότερο εμπεριστατωμένα μαζί σας. Για την Επιτροπή Προϋπολογισμών το λόγο έχει για δύο λεπτά ο συνάλφος κύριος Ντοσάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου πρώτα-πρώτα να στραφώ προς τους ε, συγγητές. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή η δουλειά τους. Και η Επιτροπή των Προπολογισμών ενέκρινε αυτό το κείμενο με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ για την συνεργασία που είχατε με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών εσείς ε, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για όλους και με αυτό το πρόγραμμα, κύριε Έτιγκερ, πρόκειται να θωρακίσετε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτό ο πάγιο διάλογο με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή των προπολογισμών. Το πρόγραμμα φυσκάλη αποσκοπεί σε αυτό. Στο να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Εργών των κρατών μελών και να υπάρχει τέτοιου είδου συνεργασία, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών που είναι πάρα πολύ σημαντικό ούτω ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ε, φοροδιαφυγή και να σταματήσει και το ξέπλυμα του χρήματο. Και ε, εμεί κατεβάζουμε κάποιε τροπολογίε ω πολιτική ομάδα και κινηθήκαμε σε κάποιου ε, άξονες, σε κάποια θέματα. Πρώτα-πρώτα τι γίνεται με τους ε, εμπειρογνώμονες, να υπάρχει ισότητα μεταξύ των φύλων, να ισχύσουν τα όσα προβλέπει ο ΙΕ, μιλώ για το σημείο 5, και επίσης να έχουμε και διάφορα μέτρα συνοδευτικά, να υπάρξει το πρόγραμμα κατά της απάτης, ενιαίο πρόγραμμα, και έτσι να υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις διαφορετικές για να έχουμε εξοικονομήσεις και αποτελεσματικότητα. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να φτάσουμε στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. 300 Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτό και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ε, αρκετή πλειοψηφία και έτσι τα Υπουργεία Οικονομικών, οι φορολογικέ υπηρεσίε να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικέ και έτσι να έχουμε ό,τι πόρου ε, χρειαζόμαστε να του ε, χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Μιλώ για ανθρώπινου, για οικονομικού πόρου, για τεχνικού και θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία μα με κρατών μέλλον, και έτσι ε, επίση να μπει ένα τέλο στην ομοφωνία. Γιατί η ομοφωνία στη φορολογική πολιτική έχει μια μεγάλη διαδρομή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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο θα μιλήσω υπέρ του προγράμματος ε, Φυσκάλη, γιατί είναι το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που απευθύνεται άμεσα στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά και χρηματοδοτεί τις απαραίτητες υποδομές για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών. Όσον αφορά τα έσοδα, τους φόρους, το πρόγραμμα αυτό καταφέρνει να ανταλλάσσουν εμπειρίες ε, οι εκπρόσωποι φορολογικών αρχών για να υποφεληθούν από τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα Φισκάλης είναι ανοιχτό στη συνεργασία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τρίτες χώρες υποψήφιες προς ένταξη Και αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή και την φορολογική απάτη, είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε το πρόγραμμα αυτό σε πρόσβαση από εμπειρογνώμονες τρίτων χωρών. Κατά την τωρινή ε, προγραμματική περίοδο, το πρόγραμμα Φισκάλης λειτουργεί χωρίς πρόγραμμα και πρέπει να το διατηρήσουμε και στο μέλλον. και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Φισκάλη, το οποίο θα υποβληθεί σε ψηφοφορία αύριο για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει τη δυνατότητα διευκόλυνση τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα τη φορολογία. Μετά τα διάφορα φορολογικά σκάνδαλα τα οποία είδαμε τα τελευταία χρόνια, είναι απολύτω απαραίτητο να μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα που διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ κρατών μελών για να καταπολεμήσουμε καλύτερα τη φοροδιαφυγή. Ο προπολογισμό αυτού του προγράμματο θα δοθεί κυρίω για τη βελτίωση τη υποδομή πληροφορική αλλά και στη φορολογική συνεργασία, δημιουργώντα ένα δίκτυο συνεργασία που θα επιτρέπει στι εθνικέ φορολογικέ αρχέ να ανταλλάσσουν εμπειρίε με ασφάλεια. Και όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, ως σοσιαλιστική ομάδα είμαστε υπερήφανοι που ε, καταφέραμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και την ε, κατάρτιση των ε, υπηρεσιών και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος γιατί τα παράνομα κανάλια έχουν όλα τα εργαλεία τα οποία θα τους βοηθήσουν στη φορά φοροδιαφύγη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Σβέν Γκίγκολτ. Σε ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει ο κύριο Πακέ για ένα λεπτό. Uh, Όσον ε, αφορά το πρόγραμμα Φισκάλης, πρόκειται για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε 30 φορολογικές αρχές. Η καλή συνεργασία ανάμεσα ε, στις φορολογικές αρχές είναι πολύ καλή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Φλάνδρα. Ε, το Φισκάλης είναι ένα πρόγραμμα εράσμους για τους φοροτεχνικούς. Το νυν πρόγραμμα τρέχει μέχρι το 2020 και τώρα πρόκειται μια πρόταση για την περίοδο μετά το 2020. Όμως ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτήν προβλέπεται μία αύξηση κατά 20% αν συμπεριλάβουμε και το Brexit και το Κοινοβούλιο θέλει να προσθέσει άλλο ένα 11%. Οι προτεραιότητες σε αυτό το κείμενο είναι αριστερής έμπνευση και εμεί δεν συμφωνούμε. Ε, το να εστιάσει κανείς κυρίως σε χώρες ε, του τρίτου κόσμου, αυτό δεν γίνεται. Εμείς θα θέλαμε να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στην απλούστευση, τη γραφειοκρατική, να μην υπάρχουν περισσότερες εκθέσεις και έλεγχοι. Ελπίζουμε να υπάρξει βελτίωση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Και ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Προχωρούμε με τον κύριο Ροζάτη για 1,5 λεπτό. Yes, thank you, thank you, President, uh, Commissioner. One of this parliament... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι βασική προτεραιότητα του πρωτοβουλίου για αυτή τη θητεία που ολοκληρώνεται όπου να είναι η καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, φορολογικής απάτης, αλλά ε, έχουμε εξεργαστεί το θέμα διάφορες ε, επιτροπές. Και το θέμα είναι η συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων αυτή η συνεργασία, δεν ήταν γνώμη των φαινομένων αυτών τόσο αποτελεσματική. Οπότε το πρόγραμμα Ευησκάλης είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και η έκθεση αυτή είναι αξιόλογη και συγχαρητήρια προ τον Σιβέν Γκίγκολ. Δυστυχώ δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Αλλά μπράβο και στην κυρία Σκοτ Κέιτο για την βοήθειά της, τη συμβολή τη που ήταν πολύ σημαντική. Εγώ να πω ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόβλημα το τεχνικό, να υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία οι επιμέρους αρχές, οι εθνικές αρχές να ε, ανταλλάσσουν τεχνολογίες και μόνο έτσι το πρόγραμμα αυτό, η ιδέα αυτή θα πετύχει. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι πολύ υπέρ αυτού του προγράμματος. Και επίσης η χρηματοδότηση θέλω να αυξηθεί, να πάει στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό είναι το ελάχιστο απαιτούμενο τόσο ώστε να έχει αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Και μην ξεχνάτε τι είδους ε, ωφελήματα μπορεί να προκύψουν γιατί είναι δισεκατομμύρια αυτά τα οποία χάνονται από την φοροδιαφυγή. Άρα το τίμημα δεν είναι τόσο μεγάλο ούτως ώστε να αναπληρώσει τις απώλειες ο κάθε κρατικός κόρβανας. Άρα ε, θεωρώ ότι η πολιτική μας πρέπει να υποστήριξει το πρόγραμμα. και για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε χρόνο εκατομμύρια φορολογικών εσόδων χάνονται ή δεν εισπράττονται γιατί υπάρχουν μορφώματα που δεν είναι και δύσκολο να δημιουργηθούν ώστε τα χρήματα να περνάνε σε φορολογικούς παραδείσους είτε μέσω του καρουσέλ στο ΦΠΑ είτε μέσω άλλων μεθόδων καταφέρνουν οι απαταιώνες να δημιουργούν συστήματα τα οποία δεν μπορούν ε, να ανακαλύψουν οι εθνικές αρχές και αυτό είναι αυξανόμενο πρόβλημα λόγω της, ε, του εξυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης. Ε, οι εταιρείε καταφέρνουν να δημιουργούν παρατήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, αποφεύγοντας την φορολόγηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εύκολο να φορολογηθούν γιατί έχουν την έδρα τους μέσα σε εθνικές ε, επικράτειες αλλά οι πολυεθνικές εταιρείες είναι πολύ δύσκολο να εποπτευθούν και γι' αυτό χρειάζεται η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι οι φορολογικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους αρκετές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν τι είναι σάπιο μέσα σε αυτό αυτό το θέμα. Αλλά ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και την περίπτωση φορολογικών ε, παραδείσων ε, και συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών ώστε να μειώσουμε τη φορολογική απάτη και να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch Έχω μόνο ένα αίτημα από τον κύριο Μαριά. Το κάνω δεκτό. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και οι φοροαπάτες βεβαίως είναι στην ημερήσια διάταξη με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία. Φυσικά υπάρχουν τα συστήματα που έχουμε δει, το καρουζέλ, υπάρχει η απάτη, αλλά άργησε η ευρωπαϊκή ένωση διότι ανέχθηκε και δεν προχώρησε στο να χτυπήσει τις φοραπάτες. είδαμε την λίστα Φαλτσιάνη, δεν είδαμε σημαντικά αποτελέσματα ανέχθηκε τα tax rulings με ιδιαίτερη ρύθμιση φορολογική στο λουξεμβούργο και στην ολλανδία. πρέπει λοιπόν να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις και να αλλάξουμε την νομοθεσία. οφείλει κάθε πολυεθνική να πληρώνει τους φόρους εκεί όπου βγάζει τα κέρδη πρέπει να κλείσουν τα διάφορα νομικά παραθυράκια γιατί έτσι γίνεται κυρίως η φοροαποφυγή και φυσικά να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών από πλευράς φορολογικών αρχών να ληφθούν μέτρα προκειμένου να χτυπηθούν οι απάτες. όμως να αλλάξουν και την νομοθεσία διότι η νομοθεσία επιτρέπει να υπάρχουν τα διάφορα νομικά παράθυρα και έτσι να φοροαποφεύγουν κυρίως οι πολυεθνικές χρησιμοποιώντας τις τριγωνικές σχέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ του Κατσδιάη. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Σέτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ε, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους περισσότερους όσον αφορά την εργασία του εισηγητή του κυρίου Γκίγκολτ και επίσης και όσον αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνέχιση του προγράμματος Φισκάλης. Ε, προτείνουμε να εκμεταλλευτούμε την καλή εμπειρία του παρελθόντος, να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ε, εσείς αναφερθήκατε στην δημοσιονομική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς προτείνουμε το ποσό των 270 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα έτη και θεωρούμε ότι το ποσό αυτό είναι επαρκές. Ε, Βεβαίω ε, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει πάντα και περισσότερα χρήματα, αλλά τα χρήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αγορά ε, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ε, λογισμικό, αλλά αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία και παίζει ρόλο είναι να καταπολεμήσουμε τις απάτες. Αυτό ενδιαφέρει όλες τις φορολογικές αρχές. Ενδιαφέρει να συνεχιστεί ο αγώνας κατά των φορολογικών αποτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Το λόγο έχει η κυρία Σκοτ Κάτω για δύο λεπτά εξ ονόματος του εισηγητή, κύριου Γκίκολτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο στο να συζητήσουμε το άρθρο 116 και καταλαβαίνω τα προβλήματα στο να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Αλλά θα ήθελα να πω, επειδή το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα φορολογικά θέματα, απογοητευόμαστε με την πολύ αργή πρόοδο και πιστεύω ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, του οποίου εκπροσωπούμε, αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε και τα πλούσια άτομα πληρώνουν του φόρου του. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουν τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο τη παρούσα συζήτηση, μου δόθηκε έπαινος για πολύ ε, λίγη δουλειά που έκανα. Όλη αυτή την εκτίμηση και τον, τους επένους θα τους μεταφέρω στον Σβέν. Ξέρω ότι και εκείνο ε, ευχαριστεί όλου του συναδέλφου για την εξαιρετική δουλειά που έγινε και για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Ελπίζουμε ότι την ίδια ευρεία υποστήριξη θα έχουμε αύριο και στην ψηφοφορία, ούτω ώστε να περάσουμε στι διοργανικέ διαπραγματεύσει την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίω και θα μεταφέρω τι ευχαριστίε σα στο Σβέν Κίγκολτ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Βαλέρο με θέμα τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες». Το λόγο έχει η κυρία Βαλέρο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές. Ε, θέλω να σας πω ότι ε, συνεργαστήκαμε με πάρα πολλές ε, οργανώσεις, με υπαλλήλου, με τη γραμματεία. Είναι πολύ καλό βέβαια να μπορεί κανείς να συνεργάζεται. Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν είναι να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε τις αρχές μας. Πρόκειται κυρίως για την ελευθερία ε, των απόψεων, προστασία των μειονοτήτων. Στη δημοκρατία αυτό που πρέπει να φροντίζουμε είναι να παρασπιζόμαστε τα δικαιώματα των μηνωτήτων γιατί τελείως δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία ε, υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά η δικαιοσύνη, αν δεν είναι ανεξάρτητη, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορούμε να εμπιστευόμαστε την ε, δικαιοσύνη. Ο δήμαρχος του Γκτάντσκ δέχτηκε την επίθεση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δημοκρατία ε, βρίσκεται σε δοκιμασία. Ασκείται πίεση, ασκείται πίεση και βία. Μεταξύ άλλων θεωρώ ότι θα πρέπει να εξτάσουμε και τη στάση μας ε, έναντι των προσφύγων. Σε πολλές χώρες ε, εκφράζονται ισχυρισμοί για διαφθορά, ε, υπάρχουν αιτιάσεις περί διαφθοράς και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ελεύθερη μετακίνηση. Περιορίζονται και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όλα αυτά είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός σε της ε, Μάλτας ασκείται κριτική εναντί αυτού. Ο κατάλογος είναι μακρύ, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πρόγραμμα για τις αξίε και τα δικαιώματα. Το 2018 προτείνεται το πρόγραμμα αυτό να εφαρμόζεται και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται κυρίως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σύνορα. Ε, χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομείς σε αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης ε, και ε, τα κονδύλια δεν επαρκούν για το πρόγραμμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε να αυξηθεί το ανώτατο όριο των κονδυλίων να μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες δράσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συμβεί κάτι τέτοιο για την ε, συνεργασία. Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι θεμελιώδεις οργανώσεις. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά και η ισότητα των δύο φύλων, η συμμετοχή των πολιτών, η κατάργηση των διακρίσεων, gender mainstreaming, όλα αυτά είναι λέξεις κλειδί και γι' αυτό πρέπει να έχουμε περισσότερα κονδύλια, να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους αυτούς τους τομείς στο πρόγραμμά μας και από κοινού να αντιμετωπίσουμε την βία και την εγκληματικότητα. Σημαντικό να αυξηθούν τα κονδύλια σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό που επίσης παίζει ρόλο είναι οι κοινωνίες των πολιτών, οι κοινότητες, όλοι αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει ως εκ τούτου ε, να ε, υιοθετήσει και άλλα προγράμματα παρήματο χάρη, ε, η αύξηση που ζητάμε εμείς είναι απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τις κοινέ μας αξίες. Στο άρθρο 2 ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εκεί αναφέρεται ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί εντάσσεται και ο σεβασμός έναντι των μειονοτήτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συμβίωση στην κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει ανεκτικότητα, αλληλεγγύη, ε, ίση μεταχείριση, καμένη αδιάκριση. Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η κυρία Πιετικάινεν, εξ ονόματος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων αλλά δεν την βλέπω παρούσα στην αίθουσα. Κατά συνέπεια δίνω το λόγο στην κυρία Κιγιόμ για ένα λεπτό από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα ανόδου της μυσαλλοδοξίας και λαϊκιστικών κινημάτων και αυτό αμφισβητεί την αίσθηση του ανήκειν σε ένα κοινό χώρο. Για να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα δίνοντάς τους ένα αντίστοιχο προϋπολογισμό. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδης εισηγητής για ένα αισιόδοξο πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες για την περίοδο 21 έως 27 προτείνονται ε, κονδύλια τα οποία θα δοθούν σε τοπικές οργανώσεις και σε ομάδες πολιτών που θα δημιουργήσουν μια συμμετοχική κοινωνία συνεχίζοντας ε, ε, τη δουλειά για να δημιουργήσουμε το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι αποφασιστικό για έργα τα οποία προέρχονται από τους πολίτες, από τη βάση, από δίκτυα πόλεων ή από αδελφοποίηση πόλεων. Όλα αυτά τα έργα βοηθούν στο να δημιουργηθεί μια Ευρώπη ανοιχτή στην πολυμορφία και την πολιτιστική πολυμορφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο Γκυγιόμ και τώρα για την Ευρωπαϊκή Ετροπή και το λόγο η Επίτροπος Γιούροβα. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ήρθε η ώρα που οι κοινωνίε έχουν να αντιμετωπίσουν τον εξτρεμισμό, την ζωσπαστικοποίηση, τις διχασμούς. Ε, οπότε θα πρέπει τώρα να έχουμε ως προτεραιότητα την δικαιοσύνη και την προαγωγή των βασικών μας αξιών. Γι' αυτό και προτείνουμε για τη θέσπιση αυτού του προγράμματος δικαιωματική αξία και ο στόχος του είναι να βοηθήσει κάποιες κοινωνίες ε, ανοιχτές χωρίς αποκλεισμούς, οπότε έχουμε πρόγραμμα και για την ε, δικαιοσύνη εκτός από το συζητούμενο. Θα πρέπει να δοθεί εντολή για τις μέλους διαπραγματεύσεις, οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά δείχνει το πόσο θέλει αυτές οι αξίες να προστατευτούν, ότι θα πρέπει να τα πρόοδου με τις διαπραγματεύσεις και εμείς είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Το νέο πρόγραμμα πρόκειται να συνεχίσει να ε, χρηματοδοτεί την ισότητα των φύλων, ε, την αντιμετώπιση των ζημιών διακρίσεων, του δικαιωματών ανήλικων, ε, προστασία των γυναικών από τη βία, καταπολέμηση του ρατσισμού και άλλες τέτοιες προτεραιότητες και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα επομένω έτσι η Ευρώπη για τους Ευρωπαίους. Θα υπάρξουν ένα σωρό διάφορα επιμέρους έργα και με αυτό το νέο πρόγραμμα θα ενθαρρύνουμε και θα διευκολύνουμε την ε, ενεργή συμμετοχή, ούτως ώστε να είναι πιο δημοκρατική η Ένωση, Ένωση Δικαιωμάτων και Αξιών. Και συμφωνούμε με τις ε, απόψεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της όσον αφορά ε, την προώθηση και την θωράκιση αξιών και δικαιωμάτων. Και αυτό είναι προτεραιότητα ύψιστη. Οπότε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματο και ταυτόχρονα το πρόγραμμα δικαιώματα και να συνεχίσει να υποστηρίζει χρηματικά διάφορου δικαιούχου πέραν των οργανώσεων ε, τη ε, κοινωνία των πολιτών, διάφορου φορεί, ε, εμπειρογνώμονε, την κρατική διοίκηση, τοπικέ αρχές, μουσεία, πανεπιστήμια κλπ. Χρειάζεται μια ισορροπία να υπάρξει αυτή η πολυμορφία και ποικιλία στο πρόγραμμα το οποίο επίσης συνδέεται με το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη και γενικότερα με τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου. Εμείς πάρα πολύ προσεκτικά ε, το θεσπίσαμε, το σχεδιάσαμε, το συνέχουμε έχουμε συνέργεια, να μην έχουμε επικαλύψεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πρικοδότηση. Ποτέ δεν φτάνουν τα χρήματα, ποτέ δεν είναι αρκετά. Οπότε ε, δυστυχώ έχουμε λιγότερα χρήματα για περισσότερε προτεραιότητες. Πάντως για τα προγράμματα που σας ανέφερε και των οποίων τους στόχους ε, εξήγησα είναι εδώ να έχουμε συνδυασμό ε, των επιμέρους πόρων μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για την ε, κοινωνική ολοκλήρωση και κοινωνική ένταξη, το νέο πρόγραμμα Horizon, πόροι για έρευνα συλλογή δεδομένων, ό,τι έχει σχέση με το πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες που συζητήσαμε. Οπότε, έτσι, ακόμα και με λιγότερα χρήματα μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα. Για την Νομική Επιτροπή. Το ρόλο έχει η κυρία Κάουφμαν για ένα λεπτό. Δεν παρίσταται. Ε, καλά. Ε, ε, όταν έλθει θα μιλήσει. Και τώρα πολιτικές ομάδες. ΕΛΚ. Μπόνι. 1,5 λεπτό. Ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ήταν μεγάλη η επιτυχία μας. Τριπλασιάσαμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Δύο δις Υπάρχει για τα δικαιώματα επί τούτου πυλώνας και 850 εκατομμύρια για τους τοπικούς φορείς και πρόκειται για κάποια χρηματοδότηση που θα δίνεται με απλή διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατία. Έχουμε τώρα διατάξεις όσον αφορά τα σημεία επαφής και η βασική μας αρχή εδώ είναι η αμεροληψία. Εάν οι κυβερνήσεις είναι εχθρικές προς τις ε, κυβερνήσεις, ε, σύγχρονα οι κυβερνήσεις είναι εχθρικές προς τους φορείς της κοινωνίας, τότε δεν θα έχουν χρήματα και έχουμε αυτό το 5% αποθεματικό για τις ΜΚΟ. Όποτε έχουμε απειλή προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, θέλουμε να κυριαρχήσει ο δημοκρατικός διάλογος. Ιδίω με εκείνους που έχουν διαφορετικές απόψεις και έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Βάση είναι η συμμετοχή των πολιτών. Αποφυγή διακρίσεων. Ισχύς του κράτους δικαίου. Αυτά είναι τα θεμέλια της δημοκρατίας. Και έτσι θα καταφέρουμε να θωρακίσουμε τις κοινωνίες μας, γιατί αυτή είναι η απάντηση όποτε έχουμε το φαινόμενο κάποιων ε, κρατών μελών που θέλουν να πάνε προς τον αυταρχισμό. Και τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία Κέγγε, 1,5 λεπτό. Σεσίλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το να επενδύει κανεί στα δικαιώματα και τις αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στου πολίτε και στην ισότητα, αυτό σημαίνει να επενδύει κανεί στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει να προχωράμε στο θέμα της ε, υπηκότητας. Σημαίνει επίσης ε, να θελήσει κανείς να υπάρχει ένα περαιτέρω εργαλείο για να προχωρήσουν οι αγώνες μας κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, ε, την παρακίνηση στο μίσος, τη βία κατά των γυναικών, τον εξτρεμισμό. Μια Ευρώπη χωρίς περιορισμούς και χωρίς αποκλεισμούς τώρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο το να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις και το μίσος ε, τα οποία τροφοδοτούνται από ένα βίο πολιτικό κλίμα. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι μας ότι οι ανοιχτές κοινωνίες, οι δημοκρατικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς δεν αυτοχρηματοδοτούνται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς προτείνουμε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος έτσι ώστε να μπορούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να στηρίξουν εκείνες τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στο να υπάρχουν κοινωνικές, δημοκρατικές κοινωνίες με δικαιώματα για όλους τους πολίτες. Επενδύουμε στο μέλλον των να υπάρχει ποικιλομορφία, ε, αξίες οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ε, και εκ μέρους τώρα των ε, συντηρητικών, ο κύριος Γιούρεκ για ένα λεπτό. Παρακαλώ Μάρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ευρωπαϊκές αξίες γιατί ο κύριος Μπόνι μίλησε για ευρωπαϊκές αξίες, για τον πολιτισμό, για την καταπολέμηση της ε, ξενοφοβίας, ομοφοβίας ε, και άλλων μορφών μυσαλλοδοξίας. Πολλά λόγια για όλα αυτά, αλλά κανείς δεν μιλά για το μίσος κατά των χριστιανών. Αν δείτε τι συνέβη το 2017, είχαμε πολλά παραδείγματα μίσους κατά των χριστιανών. Το συζητούσαμε και προηγουμένω και το ανέφερα όταν μιλούσαμε για την ετήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η τροπολογία 20, την παράγραφο 11, αφορά το μίσος κατά των μουσουλμάνων. Δεν αναφέρεται όμως το μίσος κατά των χριστιανών. Δεν αναφέρεται η περιφρόνηση της πολιτιστικής μας και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Κανείς δεν υπερασπίζεται τη θρησκευτική μας κληρονομιά. Με ανησυχεί πάρα πολύ ότι το μέσο αυτό θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δημοκρατία ανελεύθερη όπως αυτή που αναφέρει ο κύριος Ορμπάν της Ευρώπης των Ελευθεριών, ο κ. Λαντσίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε έχει σημαντικούς στόχους όπως τον σεβασμό της αξιοπρέπειας, της ισότητας, ε, του περιβάλλοντος ε, είναι πολύ ευγενή αυτή η ιδέα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ αμφισημίε ε, που χαρακτηρίζουν και την Ένωση που εκπροσωπούμε. Υπάρχουν αντιφάσεις ε, που εμφανίστηκαν τους τελευταίου μήνε πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Αναλύοντα λοιπόν αυτή την πρόταση, διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη ε, κατ' ουσίαν βρίσκεται σε δημοπρασία και όποιος προσφέρει τα περισσότερα κερδίζει. Ε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο, ε, για το οποίο δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει αποδώσει την ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε τις ε, ΜΚΟ που δεν έχουν στηριχθεί επαρκώς. Αυτές βέβαια έδειξαν μία έπαρση. Υπάρχει μία τελευταία περίπτωση όπου βλέπουμε ότι εκεί διευκολύνθηκε το ε, λαθρεμπόριο ανθρώπινων όντων. Αυτές οι εξής όμως δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν ηθικοί κίνδυνοι και αυτό δεν μπορεί πια να το επιτρέπει το Κοινοβούλιο. Ο συνάδελφος κ. Σόσνιερτς για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το κείμενο και σε αυτή την οδηγία γίνεται λόγος για αντιφατικές αξίες. Δεν μπορούμε να έχουμε ελευθερία και ισότητα σε ένα και μόνο έγγραφο, γιατί αυτές είναι αντιφατικές αξίες. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικές δεξιότητες, αλλά και αξίες. Και αυτό προκαλεί την ανισότητα. Την ισότητα μπορεί κανείς να την πετύχει μόνο σε ένα ε, στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ε, τι θέλουμε, ελευθερία ή ισότητα. Ελευθερία λόγου, αυτό επιθυμούμε. Εχθές ε, εντείνατε τις κυρώσεις κατά των μελών εδώ του Κοινοβουλίου που τοποθετήθηκαν. Τι θέλετε, ελευθερία για όλους ή για εσάς. Θέλετε τη δημοκρατία, αλλά απορρίπτετε τις μπλε κάρτες. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συμμετέχουν ε, σε αυτό το μόνο στοιχείο που είναι ελεύθερο στη συζήτηση, δηλαδή η μπλε κάρτα. Πολλοί δεν θέλουν πια να δεχτούν ε, μπλε κάρτα από μένα. Εσείς αυτή τη δημοκρατία καταλαβαίνετε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κουντρίτσκα για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Κουντρίτσκα, Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν θα μπορούσε να μαντέψει ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε τις βασικές μας αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο λαϊκισμός καταστρέφει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό όντως χρειαζόμαστε μια τέτοια πρόταση για τις αξίες. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τριπλασιάζει το ποσό και αυτό είναι θετικό. Δεν είναι υπερβολικό το ποσό, διότι οι στόχοι αυτοί είναι πήγοντες. Αυτό το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες είναι συμπληρωματικό προς ε, το μηχανισμό του κράτους δικαίου. Το άρθρο 7 μιλά για τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, αλλά το πρόγραμμα αυτό αφορά την πρόληψη. Δεν είναι μια εφάπαξ λύση, είναι μια συστημική λύση που ενισχύει την κοινωνία των πολιτών ως ε, υπόβαθρο της δημοκρατίας. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Πολωνία, η κοινωνία των πολιτών είναι πολύ ενεργή και γι' αυτό προς το παρόν επιβιώνει η δημοκρατία. Αυτό το πρόγραμμα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τις αξίες μας. Ευχαριστούμε κυρία Κουντρίτσκα. Λόπες Αγγιλάρ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Κύριε Γιώργο. Λέω ότι τώρα αμφισβητείται όσο ποτέ στι θεμελιώδεις της δεξίας η Ευρώπη. Αλλά κυρίως από συμπεριφορές, από συμπεριφορές που είναι κατάφορα αντιευρωπαϊκές και που σοβούν παντού. Οπότε γι' αυτό και είναι υπέρ το Κοινοβούλιο για ένα τέτοιο έγγραφο που προωθεί τέτοιες αξίες. Με τις ΜΚΟ, την κοινωνία και αυτά να είναι όλα ε, σύντονα με την Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση. Και μιλάμε και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27. Άρα, δεσμευσή μας είναι η υπεράσπιση της Ευρώπης. Τα ακούσαμε και χθε αυτά από τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Παντού επομένως να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Να την θωρακίσουμε την Ευρώπη. Έχει πραγματικούς ή φανταστικούς εχθρούς. Και δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος, γιατί έχουμε και κάποιους πραγματικούς εχθρούς. Το μίσος, τις ε, ακρότητας, την έλλειψη αλληλεγγύης. Άρα θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση πάρα πολύ δυναμική σε αυτούς τους πραγματικούς αντιπάλους. Αυτά πρεσβεύουν και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Βόιτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα ισχυρό πρόγραμμα για αξίες και δικαιώματα. Ε, το να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, αυτό σημαίνει βέβαια ότι ε, θα πρέπει ένα τέτοιο πρόγραμμα να εφαρμόζεται στην πράξη στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα επίκαιρο παράδειγμα. Ε, ένας άνθρωπος 83 ετών καταδικάστηκε ε, σε δύο χρόνια ε, σε φυλακή γιατί μίλησε, είπε κάτι το 2009. Είναι όμως άρεστος, του ακροτηρίασαν το πόδι, τώρα και το δεύτερο πόδι. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου αυτού του έτους ο άνθρωπος αυτός ήταν σε κλινική αποκατάσταση στο Βραδιμβούργο. Εκεί όμως δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα γιατί του αφήνουν την πόρτα ανοιχτή συνέχεια και αυτός δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ε, διαμαρτυρήθηκε και αυτό είναι το επίκαιρο που με ταράζει πάρα πολύ. Η διευθύντρια του σοφρονιστικού καταστήματος ε, επέτρεψε να κλείσει η πόρτα αλλά ε, έδωσε εντολή αυτό τον άνθρωπο που δεν έχει πόδια γιατί το έχουν κόψει να είναι δεμένος με αλυσίδες στο κρεβάτι και αν θέλει να πάει στην τουαλέτα ή να κάνει τίποτα άλλο πρέπει να φωνάξει τον φύλακα. αυτό τώρα τι είναι, και δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόιτ. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Επιτίδιο. Τη δέχεστε αυτή την μπλε κάρτα. Μάλιστα, τη δέχομαι την μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα διότι δεχτήκατε την ερώτησή μου, ήθελα να σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Αυτό το απαράδεκτο και απάνθρωπο περιστατικό το οποίο προσβάλλει τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό μας έχει γίνει γνωστό στον γερμανικό λαό και αν ναι με ποιο τρόπο αντιδρά αυτός. Τίποτα. Δεν μιλάνε. Ξέρετε, στη Γερμανία δεν είναι και αυτό μια μονομένη περίπτωση. Η γυναίκα ήταν αυτή, 90 ετών, ε, που συνελήφθη επειδή είπε την άποψή τη. Ε, και στη Γερμανία έχουμε πάνω από χίλιου πατριώτε εγκλισμένου λόγω ελεύθερη έκφραση απόψεων. Τα μέσα ενημέρωση δεν λένε τίποτα. Περίπου το ίδιο όπω και εσά ε, στην Ελλάδα. Και εσεί είσαστε βουλευτέ ενό κόμματο που φυλακίζονται οι βουλευτέ βουλευτέ σας παρότι το κόμμα σας εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πια αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Και τώρα ευχαριστώ για η κυρία Σόντρουβα και τον λόγο. Για 1,5 λεπτό Μικάλεξ τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Βόιτ, δεν χρειάζεται να επιστρατεύετε την σιωπή. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο γιατί επικρατεί η ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μπορεί κανείς να ε, δίνει, να απονέμει δικαιοσύνη, γιατί κάποιοι τη χρειάζονται. Αυτό σας είπαμε. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Εσείς αμφισβητείτε την αρχή της ισότητας. Μάλλον τα έχετε μπλέξει. Άλλο ισότητα και άλλο ομοιογένεια. Αν είστε χριστιανός, θα ξέρατε ότι η ισότητα είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πασχίζουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, βέβαια. Το πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Ισότητα για τους ε, Ευρωπαίους. Και αυτό θα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα. Το είπαμε στην Επιτροπή μας. Άρα, συμφωνώ ε, και με την αύξηση της πρικοδότησης. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι τόσο οικεία στον κόσμο. Ελπίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγήσει σε ποιοτικά έργα, σε ποιοτικά προγράμματα για όλους, για τις πόλεις, θα υπάρξει αδελφοποίηση πόλεων και κοινοτήτων. Αυτά θα μας κάνουν πιο πλούσια την εμπειρία. Ευχαριστώ. Κύριε Σόντρο. Μπλε κάρτα. Από τον κύριο Σόσνιωτς. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Κυρία Σόντροβα. Μάλιστα. Κύριε Σόσνιωτς, έχετε το λόγο. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Σόιντροβα, λέτε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ισότητα και ισότητα δικαιωμάτων ίσων ευκαιριών. Μα ισότητα σημαίνει ότι όλοι έχουμε τα ίδια μέσα στη διάθεσή μα. Μα αυτά που λέτε αντιφάσκουν. Τα μεν προ τα δε. Άλλοι κερδίζουν περισσότερα, ή λιγότερα. Επομένω, αν θέλετε ισότητα, θα πρέπει να πάρετε λεφτά από μερικού και να τα δώσετε στου υπόλοιπου που έχουν λιγότερα. Η κυρία Σόντριβα, μα κοιτάξτε. Σα άκουσα και σας πρόσεχα όταν μιλούσατε. Θεωρώ ότι ισότης ενώπιον του νόμου και ισότης όσον αφορά τα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουν όλοι. Είναι για όλους σημαντική η ισότητα ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα θα πρέπει βεβαίω και να αποφροντίσουμε να υπάρχουν ίσε ευκαιρίε. Ευχαριστούμε κύριε Σότερβαλίου Πρόεδρο. Και τώρα δίνει το λόγο στην κυρία Γουόρντ. Ένα λεπτό. Τζούλι. Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Αξίες ε, σήμερα είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ. Οι θεμελιώδεις αξίες πίσω από την ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Συχνά υποστηρίζω έργα της κοινωνίας των πολιτών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε τις αξίες όπως ε, ο πλουραλισμός ε, και η ισότητα. Να μην μένουμε στα λόγια, αλλά να έχουμε συγκεκριμένα έργα για να ενισχύσουμε τις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε δυστυχώς ότι ε, υπάρχει μια διάβρωση των αξιών στην Ουγγαρία, όπου παραβιάζονται οι νόμοι σχετικά με τους ε, πρόσφυγες. Οι δημοκρατικές αξίες θα πρέπει να υποστηρίζονται κυρίως από τους πολίτες. Χαιρετίζω τις τροπολογίες οι οποίες ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή ως ε, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η συμμετοχή των πολιτών ε, θα ενισχύσει τη δημοκρατική διαδικασία που είναι συνεκτικός παράγον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αρνηθούμε οποιοδήποτε αρνητισμό και να δώσουμε την αξία ε, στις ευρωπαϊκές αξίες. Η Τερέζα Μέη ψήφισε υπέρ του να βγούμε από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντροπή τη που στρέφεται κατά των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλοί σε ολόκληρο τον κόσμο ε, που ζουν κάτω από συνθήκες καταπίεσης και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα, για μισό λεπτό, παρακαλώ η Σίλβια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, α, για, τις εισηγήτρες για αυτή τη δουλειά. Θεωρούμε ότι ε, αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε τρία επίκαιρα προγράμματα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κυρία Γκυγιόμ ε, γιατί πρέπει να δράξουμε την ε, ευκαιρία της ηθαγένειας να ενταχθεί και αυτό το θέμα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει πρικοδοτηθεί με ειδικά κονδύλια που να αφορούν τους Φοιτητέ, ε, της αδελφοποίησης των πόλεων. Όλα αυτά πρέπει κάπως να ενταχθούν μέσα σε αυτό το νέο πρόγραμμα, ε, το οποίο είναι ένα αναδυόμενο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που ήταν η Ευρώπη των πολιτών και τώρα βρίσκεται μέσα στο δικό μας το πρόγραμμα να παραμείνει συνδεδεμένο ε, με την μνήμη την οποία πρέπει να συμμεριζόμαστε όλοι μια ιστορική μνήμη η δυνατότητα να έχουμε μια μια κοινή ιστορία και από την άλλη οι πολίτες να κατανοούν ότι θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε μια νέα Ευρώπη. Αγώνας κατά του ρατσισμού, του μίσους, ε, των διαφόρων μορφών του εθνικισμού ε, που διαπνέουν την Ευρώπη. Ε, το θέμα της ηθαγένειας είναι ένα θέμα ουσιαστικό και γι' αυτό πρέπει να εκταμιευτούν επιπρόσθετα κονδύλια, να υπάρχουν αρμοδιότητες για την ηθαγένεια, ακόμα και μέσα από άτυπη και ε, τυπική εκπαίδευση. Ε, εμείς ε, θελήσαμε να εντάξουμε και το θέμα του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου γιατί πρέπει να υπάρχει μια κοινή προοπτική της ευρωπαϊκής σίνης. Τώρα λοιπόν διαδικασία Catch the Eye. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. <clears throat> Θα δεχτώ και τις δύο. από τον κύριο τον Ακούραστο, τον κύριο Μαριά ξεκινάω. Κύριε Μαριά ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα θα δοθεί για τη στήριξη των αξιών της ένωσης 474 εκατομμύρια για την ισότητα και τα δικαιώματα 500 εκατομμύρια για τη δραστηριοποίηση των πολιτών όλα αυτά με στόχο να ενισχυθούν οι ίδιοι οι πολίτες. θεωρώ ότι η καλύτερη στήριξη για τους πολίτες είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για εργασία διότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει αξιοπρέπεια. Και την εργασία η ευρωπαϊκή ένωση στο θέμα το γνωστό για την εγγύηση για την νεολαία έχει δώσει μόνο έξι δισεκατομμύρια. εγώ βλέπω ότι το ποσό το οποίο θα διατεθεί δύο δισεκατομμύρια στις ΜΚΟ θα δώσει ευκαιρία σε πολλές ΜΚΟ να κάνουν το γνωστό πάρτι ό,τι έκαναν και με τα κονδύλια που δόθηκαν για τη μετανάστευση. γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει προσοχή. από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα κονδύλια πρέπει να πάνε στα πανεπιστήμια στα σχολεία στους δήμους στις περιφέρειες και φυσικά να δοθούν για την αντιμετώπιση του μίσους κατά των χριστιανών. να επισημάνω ότι υπάρχουν το 2017 έγιναν 556 επιθέσεις στην ελλάδα το 94% κατά της ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας. θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μην είναι μονομερές. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Κύριε για ένα λεπτό. Ε, σε μια εποχή κατά την οποία όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υφίστανται οικονομικά προβλήματα και οι λαοί τους υποφέρουν, ο ηγετικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισε να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Δικαιώματα και Αξίες. Στην έκθεση γίνονται προτάσεις για να διατεθούν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να προαχθούν και να προστατευτούν η δημοκρατία η ισότητα το κράτος δικαίου και να αντιμετωπιστούν όλες οι μορφές της βίας. κάποιος όμως πρέπει να επισημάνει σε αυτούς τους πεφωτισμένους εγκεφάλους της ευρωπαϊκής ενώσεως ότι η δημοκρατία η αγάπη προς την ισότητα τις αξίες ο σεβασμός των πάσης φύσεως δικαιωμάτων είναι αποτέλεσμα συνειδήσεως και πνευματικής καλλιέργειας και όχι αντικείμενο μιας κερδοσκοπικής επιχειρήσεως. ως εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού θεωρώ ότι δεν έχω το δικαίωμα να ανεχθώ να... και να συνενέσω να ελοποιηθεί αυτό το όργιο κατασπαταλήσεως των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων από την ευρωπαϊκή ένωση η οποία έχει καταδικάσει του συμπατριώτες μου σε λιτότητα και εξαθλίωση. γι' αυτό λοιπόν δεν θα υποστηρίξω την έκθεση και καλό να κάνουν το ίδιο όσες και όσοι αισθάνονται ότι έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τους τίμησαν με την ψήφο τους. Ευχαριστώ πολύ.